περιφερειών σε σχέση με το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στους αστικούς χώρους. Θέτω την πρόταση αυτή σε ψηφοφορία με ονομαστική ψήφο. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The roll call vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία, λέγω. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή η αίτηση για διαβούλευση. Κύριε Πρόεδρε, χθε άφησα εδώ την κάρτα ψηφοφορίας μου. Αλλά όταν ήρθα σήμερα είδα να απουσιάζει η κάρτα μου. Γι' αυτό δεν έχω κάρτα, ούτε δύναμη καν να ψηφίσω, όπως θα όφυλα. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να ελέγξουν πού ετέθη η κάρτα μου, πού έχουν πάρει την κάρτα μου. υπάρχουν πάντα κάρτες αντικατάστασης από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Φοβάμαι ότι αυτό θα πρέπει να πράξετε. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η ψηφοφορία βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας της εκθέσεως του κυρίου Όνεστα και δίνω το λόγο στον κύριο Κρόουλη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που διακόπτω την ψηφοφορία, αλλά βάσει του άρθρου 170 του κανονισμού μας ζητώ την αναβολή της ψηφοφορίας για την έκθεση όνεστα σε σχέση με τη διαδικασία αναφορών. Γιατί το θέμα αυτό είναι υποσυζήτηση στη συνέλευση των Προέδρων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα αυτό των μεταρρυθμίσεων που αυτόνται τι εκθέσει όνεστα θα συζητηθεί στι 5 Μαρτίου και επομένως ζητώ μέχρι τότε να αναβληθεί η ψηφοφορία και να εξεταστεί στη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου στην Σύνοδο του Στρασβούργου. Ευχαριστώ κύριε Κρόουλη. Ένας ομιλητής υπέρ και ένας κατά. Ο κύριος Ωνεστά, ναι, κύριε Πρόεδρε. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η έκθεση αυτή τροποποιεί τον κανονισμό μας ή τον αποσαφηνίζει καλύτερα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι αναφορές της Επιτροπής Αναφορών αν θεωρούνται παραδεκτές, δεν θεωρούνται παραδεκτές, τι πληροφορίες δίνουμε στους αναφερόμενους κτλ. Ενεκρίθη στην Συνταγματική Επιτροπή με ομοφωνία μείον μία ψήφο. Δεν είναι αφιλεγόμενη λοιπόν αυτή η έκθεση, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο όπου αποφασίσαμε να διευκρινίσουμε ότι όταν τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας, αν τεθεί σε εφαρμογή, τότε οι αναφορές που έχουν να κάνουν όχι με το Κοινοβούλιο αλλά με την Κομισιόν, στην Κομισιόν, πρόκειται για λαϊκές πρωτοβουλίες με ένα εκατομμύριο υπογραφές, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει απλώς να αναφέρεται αυτό στον, ε, στους αναφερόμενους. Αυτό είναι όμως σε μια υποθετική κατάσταση. Εγώ μπορώ να δεχτώ την ε, καθυστέρηση μέχρι τις 5 Μαρτίου, ακόμα και μια τροπολογία που θα αφαιρέσει αυτό το στοιχείο. Αλλά θα είναι, ε, θα είναι λανθασμένο να αλλάξουμε τον κανονισμό μας δημιουργώντας προβλήματα στο μέλλον. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Όχι, οπότε τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της αναβολής παρακαλώ. Ευχαριστώ αυτή μου κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η αναβολή της, ε, εκθέσης, της εξαίρεσης εκθέσης εκθεσης εκθεσεις εξαιρεσης ακολουθούμε με την ψηφοφορία βάσει της απλοποιημένης πάλι διαδικασία της έκθεσης της κυρίας Ριέρα Μαδουρέλ για την Ευρωπαϊκή Υποδομή Έρευνας. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. Συγχαρητήρια στην κυρία Μαδουρέλ. Ακολουθεί η ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Μόρι Γιόν βάσει απλοποιημένη διαδικασίε σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση για Πολυμερή Συνεργασία στον Βορειοατλαντικό Αλληλευτικό Χώρο. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη στρατηγία Μοριών. Ακολουθεί η έκθεση Κίνοκ για την ειδικό χώρο για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Εξωτερική Δράση, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Κίνοκ. Ακολουθεί η ψηφοφορία της έκθεσης του, κυρίου Κοτινή για το Γενικό Πλαίσιο Πληροφόρησης και διαβούλευση με τους εργαζομένους. Ονομαστική κλίση, άρχιδη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια στην εισηγητή. Ακολουθεί η έκθεση της κυρίας Τόγια για την κοινωνική οικονομία. Η εισηγήτρια θέλει να προτείνει μια προφορική τροποποίηση σε ένα σημείο της ε, έκθεσης. Κυρία Τόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω στην παράγραφο 12 πριν μιλήσουμε για την κοινωνική οικονομία να βάζουμε και την λέξη components συστατικά. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Τίθεται σε ψηφοφορία, τροπολογημένη, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Δεκτή. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Σαμπάζη για την ψυχική ηχεία Ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Γιώργκ για τα εθνικά προγράμματα δράσης στον τομέα της αποτελεσματικότητας τη ενέργειας. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος τη ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Ράμος για την εφαρμοσμένη έρευνα σε σχέση με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ονομαστική. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Συγχαρητήρια στην κυρία Ράμος. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Σέντερσολτ για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα για τους παροχείς υπηρεσιών. Πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Σέντερ Σολέχτια το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήταν σημαντικό να ξέρουμε πόσο ικανοποιημένοι θα ήταν όλοι αν δεν μιλούσα για δύο λεπτά. Θα περιοριστώ λοιπόν να πω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς επανειλημμένα προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τη ζωή των πολιτών μας, να τους κάνουμε πιο εύκολο να <clears throat> ξεκινήσουν μια επαγγελματική δραστηριότητα διαμεθοριακού χαρακτήρα. Αυτό είναι σημαντικό για την εκλογική εκστρατεία ενόψη των εκλογών και θα το αναφέρω μονάχα έτσι, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ κυρία Σέντερσον. Ονομαστική κλίση για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Σέντερ Σόλτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά σας αναφέρω ότι υποδεχόμαστε σήμερα μια αντιπροσωπεία βουλευτών και άλλων επισκεφτών από την πολιτεία των μεγάλων ουραλίων από τη Μογγολία και επίσης καλεσμένους από την αποστολή της Μογγολίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βρίσκονται στα επίσημα θεωρία.